So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Καλημέρα, αγαπητοί φίλοι. Και συνάδελφοι, μπορούμε να συνεχίσουμε στην ημερήσια διάταξη. Με το σημείο 6. θέση του Κοινοβουλίου για το σχέδιο προπολογισμού του 2011, όπω το έχει τροποποιηθεί από, την Ευρωπαϊ... από το Συμβούλιο. Και εδώ έχουμε τροπολογίες από την Επιτροπή μας. Η κυρία Γιούτα Χάουκ δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Η συγγήτρια, η συντάκτης. Θα ακούσουμε λοιπόν την κυρία Λίντα Μακέδων, η οποία θα μας πει τι ε, γνώμη έχει η Επιτροπή για τον προπολογισμό 2011. Ζητεί συγγνώμη η Ιούτα Τα ξέρει πολύ κατά θέματα του προπολογισμού από ότι εγώ. Και είπαμε να κάνουμε κάτι πριν έρθει ο νέο γύρο των διαπραγματεύσεων. Και εδώ έχει την αιτιολογημένη γνώμη τη. Και σήμερα μου ζήτησε να σας πω ότι έχουν γίνει διαπραγματεύσεις με την Γραμματεία, τη Γενική Διεύθυνση για τα Οικονομικά, για το Περιβάλλον και η ονοματολογία έχει αλλάξει γιατί έχουμε τη δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης όσον αφορά την πολιτική για το κλίμα και αν κοιτάξετε τώρα τον προϋπολογισμό και έχουμε τώρα και τις αντίστοιχες γραμμές προϋπολογισμού, τα κονδύλια. Η Γιούτα ήθελε να τονίσει αυτό το πάγιο πρόβλημα του Ταμείου για το τα είδη καπνό ε, ένα ταμείο το οποίο πρόκειται να εκπνεύσει η περίοδος ισχύου το, το 2010 Καφέ, Καφέ. Αυτά τα λέει στο σημείο 5 και λέμε ε, ότι η Γενική Διεύθυνση για, για τα Γερικά μπορεί να βρει μια λύση. Διάφοροι συνάδελφοι έχουν ε, υποβάλει πιλωτικά προγράμματα και έχουν προτείνει κάποιες δράσεις για τον προϋπολογισμό και η Επιτροπή αντέδρασε κατόπιν της δημοσίευσης του Ιουλίου και Υπενθυμίζω ότι τα πιλωτικά προγράμματα έχουν ε, πειραματικό καινοτόμο χαρακτήρα για να δοκιμαστεί αν μια δράση είναι χρήσιμη. Και είπαμε να εκπονηθούν κάποιες προτάσεις για μέλουσες δράσεις. Εννοεί, νομίζω, ότι εξετάζονται αυτά τα προγράμματα επί τη βάση αυτών των ε, ορισμών του τι είναι ε, τέτοια δράση και τέτοιο πρόγραμμα πιλωτικό. Ζητεί να εξεταστεί το χρονοδιάγραμμα 19 Εβδόμου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες και για τις ε, τροπολογίες του προπολογισμού τις έστειλε η γραμματεία στις 7 Εβδόμου την προηγούμενη εβδομάδα και θα γίνει η ψηφοφορία στις 6 ενάτου στο Στρασβούργο. Η Γιούτα λέει ότι ευχαριστεί την Γραμματεία και συγκεκριμένα την Εμίλια Ρωμάνο για τη δουλειά τη όσον αφορά την προετοιμασία του προπολογισμού. Αυτά μου ζήτησε η Γιούτα να σα πω. Πέστε μου με την παρατήρηση σας για το σχέδιο του κειμένου και θα τις θα διαβιβάσω. Ευχαριστώ για την έκθεση εκ μέρου τη Ιούτα. Η γραμματεία άκουσε ήδη τι ευχαριστίε. Σχόλια υπάρχουν. Ε, θέλει κανεί να λάβει το λόγο για το θέμα αυτό. Όχι. Από ό,τι φαίνεται, σας έχει καταλάβει όλους η κόποση. Ή αλλιώ είστε όλοι πολύ ικανοποιημένοι, μάλλον αυτό να πούμε. Καλύτερα ευχαριστημένοι παρά κουρασμένοι. Εντάξει, λοιπόν, γνωστές ημερομηνίες λάβαμε την ενημέρωση. Ε, έχουμε κάπως ε, προχωρήσει πιο γρήγορα στο θέμα των ε, ψηφοφοριών που έχουμε προβλέψει για τις 9.30. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημέρας της διάταξης. Έκθεση για την εφαρμογή των ε, προδιαγραφών για την ε, βιοπικιλότητα. Πρόκειται για την έκθεση Ντελάνγκε που φαντάζομαι έρχεται. Έχουμε 104 τροπολογίες στο θέμα αυτό. Richard. Πρόεδρε, μια και είναι για τις 9.30 η ψηφοφορία στην ημερήσια διάταξη εγγεγραμμένα ε, και είναι λίγοι συνάδελφοι εδώ. Μήπως να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα μέχρι ότου συγκεντρωθούμε όλοι. Αφού το λέει η ημερήσια διάταξη, θα συγκεντρωθούμε, ξεκινήσουμε στις 9.30. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Θα έλεγα τότε να δούμε την έκθεση για την αντιπροσωπεία μας στην ΕΦΣΑ, στο σημείο 11 της ημερησίας διάταξης. Να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Όπως έλεγα λοιπόν, είχαμε πάει στην ε, Πάρμα. Επτά ε, μέλη είχε η αντιπροσωπεία μας, την έκθεση την είδατε. Η ΕΦΣΑ, ξέρετε, είναι αυτή η αποκεντρωμένη υπηρεσία η οποία ισχύει, ε, άρχισε να λειτουργεί από το 2002 και ύστερα από τα ε, διατροφικά σκάνδαλα που γνωρίσαμε στη δεκαετία του 2000. Έχει καθήκον να καταθέτει ανεξάρτητες εκθέσεις ε, για ζητήματα που αφορούν τη διατροφική αλυσίδα. Με τον κύριο Νταλίχ, η συζήτηση μάλιστα έθιξε και το ζήτημα της αξιολόγησης κινδύνου στην οποία προβαίνει η ΕΦΣΑ Ακούστηκαν κάποιε αιτιάσει από πλευρά της δική μα ε, πλευράς ως προς την ποιότητα των ε, επιστημόνων, ε, δηλαδή την κατάρτισή τους, την ανεξαρτησία τους, αλλά και την κατάρτιση επιστημονικών εκθέσεων που καλύπτουν ή πρέπει να καλύπτουν διαφορετικά θέματα. Η ΕΦΣΑ είναι μια υπηρεσία σε ανάπτυξη αυτή τη στιγμή. Ξέρετε την ιστορία του, της έδρας, την περίφημη ιστορία της έδρας, την Πάρμα. Ξέρετε ότι δεν επελήθη πολύ εύκολα αυτή η υπόθεση. Και τι έχει προχωρήσει σε βελτίωση η υπόθεση, γιατί εξασφαλίζεται νέο ε, κτίριο για την ΕΦΣΑ και για τους υπαλλήλου της, οικογένειας με παιδιά ιδιαίτερα που έχουν ε, ανάγκη. Προβλέπεται και η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού σχολείου, ώστε να μην χρειάζεται τα παιδιά τους να πηγαίνουν στην Ίσπρα, που είναι αρκετά μακριά, για να παρακολουθούν τα μαθήματα στο εκεί ευρωπαϊκό σχολείο. Συστήσαμε λοιπόν όλα τα καυτά θέματα, τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που συζητήσαμε και χτες, ε, τα νέα τρόφιμα, κλωνοποιημένο κρέας, βιοκτώνα, μπισφενόλες ένα, διφενόλες συγγνώμη και ζήτημα των ε, κινδύνων για την υγεία. Ε, ξέρετε ότι έχει, όπως έλεγα και νωρίτερα, πολλά και δύσκολα θέματα η ΕΦΣΑ ε, στις αρμοδιότητές της, αλλά και εμείς πρέπει από πλευράς μας να μεριμνούμε έτσι ώστε να μην την ε, κατηγορούμε άδικα. Ε, δεν μπορούμε σας να ισχυριστούμε λοιπόν ότι δεν είναι ανεξάρτητη η ΕΦΣΑ, αλλά ε, διαπιστώνουμε ότι δεν καταρτίζονται επαρκής, επαρκώς ε, ευάριθμες, επαρκώς ε, αρκετές εκθέσεις για τα ζητήματα που μας απασχολούν. Εν πάση περιπτώσει, ήταν καλό το ότι το Κοινοβούλιο έδειξε ενδιαφέρον για την ΕΜΣΑ. και οι ίδιοι 304, 304 ε, μέλη του προσωπικού της ΕΦΣΑ θεώρησαν ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για αυτούς και για την ανταλλαγή απόψεων βέβαια αλλά και για να παρουσιάσουν το έργο τους. Και είδαμε όπως έχουμε δει και άλλες φορές ότι οι επισκέψεις μας ε, στις αποκεντρωμένες υπηρεσίε την χάνουν ιδιαίτερης Εκτίμηση από το προσωπικό, γιατί και αυτοί μένουν και δουλεύουν μακριά από τις Βρυξέλλες και χρειάζονται την επαφή. Θέλουν λοιπόν να βλέπουν τις επισκέψεις των βουλευτών τακτικά. Είχαμε αρκετούς συναδέλφους παρόντες στην αντιπροσωπεία. Δεν ξέρω αν κάποιος από αυτούς θέλει να παρατηρήσει κάτι, αν υπάρχουν ερωτήσεις. Κύριε Ζέμπαχ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τα συμπεράσματα από την επίσκεψη καταγράφονται στην έκθεση μέσα από διάφορες επικρίσεις για την αξιολόγηση κινδύνου, παραδείγματι όπου δεν είμαστε πάντοτε ικανοποιημένοι για τα όσα μας έχει πει η ΕΦΣΑ και για τα προϊόντα κλωνοποιημένου κρέατος και για τους ιδιωτικά τροποποιημένους οργανισμούς και για τις αρωματικές ουσίες κλπ. Αλλά πιο συγκεκριμένα ε, ε, περιθώριο βελτίωσης ε, τι συγκεκριμένα δηλαδή μπορεί να κάνει η ΕΦΣΑ για να βελτιώσει τη δουλειά της αφενός αφετέρου δε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ορατότητα της υπηρεσίας και της δουλειάς της τα έχετε συζητήσει πιο αναλυτικά έχετε κάποιες συγκεκριμένε ιδέες απάντηση ναι δεν είναι οι επικρίσεις κάτι το καινούριο τις έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν και ο Επίτροπος Δαλή ο ίδιος επισκέφθηκε την ε, Πάρμα και είχαμε πει ότι μέχρι το 2010 θα πρέπει ο κανονισμός λειτουργίας της ΕΦΣΑ και όλος ο τρόπος εργασίας της να μπουν στο μικροσκόπιο. Μέχρι τα τέλη του έτου, από ό,τι μας είπα ε, χθες ο Επίτροπος, ε, θα πρέπει να υποβληθεί μια έκθεση και για τη βελτίωση, για τον τρόπο λειτουργίας, για την ανάπτυξη αυτής της, ε, για τις δομές μάλλον αυτής της αποκεντρωμένης υπηρεσίας. Και όπως είπαμε και χθες πρέπει να ενισχυθεί η φήμη της υπηρεσίας. Πρέπει να την χάνει γενικότερη αποδοχής και να είναι αποδεκτού κύρους. Όσο και αν δεν συμφωνεί κανεί ενδεχομένω με τα αποτελέσματα κάποια πραγματογνωμοσύνη, με τι πέρασματα κάποια πραγματογνωμοσύνη, οι κρίσει τη ή η ανάλυση του κινδύνου στην οποία προβαίνει, προβαίνει πρέπει να είναι και ανεξάρτητη και ποιοτική και αντικειμενική και διεξοδική. Αυτά λοιπόν θέλουμε να τα δούμε όταν έρθει η ώρα για τις μελέτες, για την επανεξέταση των μελετών της. Λίντα Μακιάβαν. Να δούμε την ερώτηση τώρα όσον αφορά αυτές τις υπηρεσίες στο γενικότερο θέμα. Αυτό που είπες Πρόεδρε, τα σχολεία και αυτοί που πρέπει να πάνε και να υπηρετήσουν, παρέχουμε. Πολλέ τέτοιε υπηρεσίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλέ από αυτέ δεν έχουν σε καθαρή εντολή και άρα θα πρέπει στο μέλλον να συγκροτούμε κάποιε υπηρεσίε μόνο εάν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που θα πρέπει να εφαρμόζεται και θα, να έχουν κάτι συγκεκριμένο να κάνουν. Να είμαστε σκληροί που με το Συμβούλιο κάθε φορά που φτιάχνουν τέτοιες υπηρεσίες σε διάφορα μέρη για να ικανοποιήσουν τον κόσμο προσλαμβάνονται κάποιοι, βρίσκονται για τους συντρόφους τους ε, κάποιες δουλειές και ε, έτσι, έτσι καθορίζεται τελικά το πώς λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες ε, ανάλογα με το ποιους βρίσκουν να δουλέψουν εκεί. Τώρα, όσον αφορά αυτές τις μελέτες ασφάλειας, να μην ξεχνούμε, ότι οι επιστήμονες απαντούν πάνω σε αυτό που Αυτό θα απαντήσουμε κάτι είναι επιστημονικά ασφαλέ και όχι αν είναι επιθυμητό κοινωνικά ή αν χρειάζεται να γίνει. Ε, Α πούμε τα κλωνοποιημένα ζώα μπορεί να είναι ασφαλέ να φας το κρέα, αλλά γιατί να θέλει η κοινωνία μα να έχει τέτοια ζώα. Λείπουν τα ζώα, τα κανονικά. Ε, δεν απαντούν σε όλα αυτά οι επιστήμονε. Μα λένε μόνο την επιστημονική του γνώμη για αυτό που του ρωτάμε. Επομένω, άλλο το να απαντούν σε κάτι και άλλο το να, να κάνουμε κι εμείς ε, ανάλογες ενέργειες. Ποτέ δεν πρόκειται να έχει κανεί όλες τις απαντήσεις πάνω στο κάτι που καίει σε κάποια συγκεκριμένη μέρα. Επομένως, ε, τα επιχειρήματα για κάτι δεν είναι πάντοτε επιστημονικά Υπάρχουν διάφορα ζητήματα όπως το καλομεταχείριση των ζώων, πούμε, για τα κλωνοποιημένα ζώα. Και αυτό ισχύει και για την ασφάλεια, για το αν κάτι είναι ασφαλέ να φαγωθεί. Για την διφενόλη α τώρα, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Ε, αν θυμάμαι καλά, κάτι πρόκειται να, να βγει από την ΕΦΣΑ ή από την ε, Κομισιόν αυτή τη βδομάδα. Κάτι θα πρόκειται να δημοσιευθεί. 13 ή 14 Ιουλίου ήταν κάτι να βγει. Καλώ Καλώς, δεν ξέρω αν από την Επιτροπή υπάρχει κανείς για να απαντήσει. Γιατί τι φαινόλες ένα. Κύριος Βόλφ. Ε. Είπαμε αυτή τη βδομάδα στο website ότι αναβάλαμε την τελική έκθεση για τα PPA για τον Σεπτέμβριο. Γιατί έχουμε 800 μελέτες να χτενίσουμε. Ja, das war die Auskunft zu Bisphenol A. Αυτέ ήταν οι πληροφορίε λοιπόν για τη διφενόλη Α, όχι τον Ιούλιο αλλά τον Σεπτέμβριο. Θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση και άλλη παρατήρηση έχει το Κοινοβούλιο καταρτήσει αρκετέ εκθέσει για τι αποκεντρωμένε υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι σχετικέ αποφάσει σε επίπεδο που λίγο πολύ επικρατεί η νοοτροπία ποιο κράτο δεν έχει υπηρεσία, να του δώσουμε μία. και όπου οι δομές επίσης, οι οργανωτικές δομές είναι πολύ διαφορετικές, έχουμε ένα ποτφουρί από οργανωτικές μορφές. Και αυτό λοιπόν θα θέλαμε και είχα και την ε, χαρά στην Επιτροπή των Σταγματικών Υποθέσεων που ήμουν πριν να παρακολουθήσω τα θέματα αυτά αρκετά συχνά. Η Λίντα λοιπόν πολύ σωστά παρατήρησε ότι όντως έχουμε συστήσει τα θέματα αυτά αρκετές φορές ε, η ΕΦΣΑ προβαίνει μόνο σε αξιολόγηση κινδύνου. Η διαχείριση του κινδύνου, δηλαδή η τελική πολιτική απόφαση ρίξει εμάς. Και όταν λαμβάνουμε τη σχετική πολιτική απόφαση, τη λαμβάνουμε όχι απαραίτητα μόνο με γνώμονα τα όσα μας είπαν οι επιστήμονες, αλλά και εκείνα τα οποία θεωρούμε πολιτικά ορθά. Αλλά βέβαια με δεδομένο ότι μετά τον διαφωτισμό επικρατεί η λογική ως κύριος γνώμονας και ως εκ τούτου προτιμούμε πάντα να στηριζόμαστε στις επιλογές μας σε επιστημονικά κριτήρια αλλά πάντως όχι αποκλειστικά ή πάντα. Το ίδιο θα ήθελα να επισημάνω για την FDA στι ΗΠΑ, ότι προβαίνει μόνο σε αξιολόγηση κινδύνου, risk assessment. Έχει καθαρά επιστημονικό χαρακτήρα, δεν έχει κοινωνικο-οικονομικές δηλαδή ε, διαπιστώσεις να αναλύσει, ενώ η ΕΦΣΑ έχει και ένα τέτοιο καθήκον, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή κάνει αξιολόγηση κινδύνου και υπό τις κοινωνικο-οικονομικές πτυχές και όχι μόνο τις επιστημονικές. Βέβαια, βαρύνουσα θέση έχει ή θα έπρεπε να έχει η επιστημονική αξιολόγηση. του ε, δε κίνδυνο, τη διαχείριση του κινδύνου θα πρέπει να την ε, κάνει ο, η Επιτροπή. Εμείς ως ε, νομοθέτες. Εν λοιπόν, τώρα ακούσαμε τα της ΕΦΣΑ. Προχωρήσαμε αρκετά καλά συζητώντας αυτό το θέμα της ημερησίας διάταξης και καλύπτοντας το χρόνο που είχαμε. Βλέπω και το Βιτόριο Πρόντι που ήταν στην, στην ε, Πάρμα. Δεν ξέρω Βιτόριο αν θες να πεις κάτι και εσύ για την ΕΦΣΑ. Αν έχεις κάποιο σχόλιο, κάτι που θέλεις να παρακατηρήσεις, Βιτόριο. Ευχαριστώ. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω όλη τη συζήτηση. Πολύ σημαντική επίσκεψη για να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια πώς ε, οργανώνονται και αντιδρούν στα μεγάλα θέματα. Η ΕΦΣΑ είναι μια οργάνωση, ένας οργανισμός βελτιώσιμος. Και μπορούμε να υπολογίζουμε σε αυτή την οργάνωση. Να στηρίξουμε την ομοθετική μας δουλειά με επαρκή γνώσεις, Δηλαδή, θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε τη λειτουργία της και να της δίνουμε κίνητρα γιατί υπάρχουν ε, θέματα όπως τα νέα τρόφιμα, οι γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί. Η πίεση επί της γεωργίας για την παραγωγή που θα δημιουργήσει νέες συνθήκες και νέες ανάγκες που πρέπει να τις παρακολουθούμε από πολύ κοντά. Πιστεύω ότι η ΕΦΣΑ μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό όργανο και για τη δική μας δουλειά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Βιτόρο και εγώ το επιβεβαιώνω. Θέλουμε βέβαια να βελτιωθούν τα αποτέλεσματα εργασία τη ΕΦΣΑ, που έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τη δική μα δουλειά. Και άρα πρέπει να μεριμνούμε και να κάνουμε την ε, κριτική μας με προσοχή και περίσκεψη. Γιατί είναι για όλα αυτά τα περίπλοκα θέματα πολύ σημαντική για μας αυτή η αποκεντρωμένη υπηρεσία. Καλώς λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα της μέρης της διάταξης ψηφοφορία της έκθεσης για την εφαρμογή της κοινωτική νομοθεσίας ως προς τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και η συγγήτρια είναι εδώ, κυρία Στερτελάνια. Είναι και αρκετοί συνάδελφοι πλέον που ήρθαν για την ψηφοφορία και ως εκ τούτου μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχετε τον κατάλογό σας. Ξεκινούμε. Τροπολογία 2.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 κατά αποχές εγκρίνεται 38 φιέλνερ σε τμήματα πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 Κυρμπράντη και λοιπή ε, σε τμήματα πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, επαληθεύουμε ηλεκτρονικά στο δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 39 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 22 κατά, 2 αποχές εγκρίνεται. Δυστυχώς. Δεν σας εξυπηρετεί το αποτέλεσμα. Έτσι γίνεται όμως. Εγκρίθηκε. Πρόεδρε, δεν έχω την κάρτα μου, δεν τη βρίσκω και όσο και δεν μπορώ να συμμετάσχω στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ναι, νομίζω ότι αν κάποιο συνάδελφο έχει φέρει την κάρτα του αλλά δεν δουλεύει, τουλάχιστον για λόγου αυρότητα, επιτρέψτε του να συμμετάσχει στην ψηφοφορία. Ε, εάν ε, κάποιο την έχει ξεχάσει και την έχει φέρει, εντάξει, αλλά κάποιο που έχει μια κάρτα που δεν δουλεύει, ε, να συμμετάσχει. Πώ το γίνει. Ε, κάρτα χαλασμένη είναι μη κάρτα. Δεν υφίσταται. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο. Καλώς λέει ο πρόεδρος. Να επαληθεύσω για άλλη μια φορά. Κοιτάξτε να σας πω, η γραμμή είναι σαφής. Γίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία στην Επιτροπή. Το γνωρίζουμε. Φέρνουμε την κάρτα μας ή δεν τη φέρνουμε γιατί την ξεχάσαμε, αλλά βάζει περιπτώσει είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι. Δεν μπορεί να έχει κανείς δικαιολογίες. Κυρία Μακάουαν αν χάλασε η κάρτα, έχουμε και μια δεύτερη κάρτα. Α στείλει η γραφείο να φέρει μια άλλη κάρτα. Έχουμε δύο ή τρει κάρτε. Μπορούσαμε να δεχτούμε τώρα, κατεξαίρεση να το δεχτούμε αυτό σήμερα. Διαφορετικά κάθε φορά θα έχουμε την ίδια συζήτηση. Και οι συνάδελφοι του είπαν ότι και αυτή τσέτυχε το ίδιο. Και πρέπει να περιμένει να έρθει η καινούργια κάρτα. Κοιτάξτε, ο κανόνας είναι σαφή. Γίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία και το αποτέλεσμά τη είναι ισχυρό. Τώρα να αρχίσω να μετράω Ποιο έφερε, ποιο δεν έφερε, ποιανού χάλασε και ποιανού δεν χάλασε, θα με επικρατήσει χάος. Αυτό μπορώ να κάνω είναι αν θέλετε για λόγου σεβασμού προ την κάρτα που χάλασε όπω λέτε να επαναλάβω την ψηφοφορία, αλλά όταν έχουμε ψηφοφορίε, πρέπει να φαίνεται τι κάρτε σα. Παραλαμβάνω λοιπόν 39 δεύτερο τμήμα. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία δεύτερο τμήμα της 39 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορίες. Μάλιστα. Πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα τώρα. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Και φαίνεται ότι θα αποδείχθη χρήσιμη η χαλασμένη κάρτα. Πάμε στη 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται, αλλά να επαληθεύσουμε αν προτιμάτε. Στη 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσαμε πέρα ψηφοφορίας 28 υπέρ, 25 κατά. Εγκρίνεται. Άξιο το κόπο για παλήθευση. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 έχει αποσυρθεί λέει ο πρόεδρος, 42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 43 καταπίπτει. Ενοποιημένη τροπολογία υπεριθμών 2 παρακαλώ τώρα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται Καταπίπτουμε σε ως κάποιες τροπολογίες και πάμε στην τροπολογία 48 ε, της παραγράφου 9 της κυρίας Μακάβων τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά άποχες. Επίσης εγκρίνεται για, το, για τη δε 53 μου λέει ο γραμματέας μας ότι έχει αποσυρθεί το πρώτο τμήμα, όχι το δεύτερο όπως λέει ο κατάλογος. Ψηφίζουμε λοιπόν το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 επαλήθευση παρακαλώ Πέρα στις φοφορίες το ΕΛΚ έχει δύο ψήφους περισσευούμενες, πρέπει να πάρει, να αφαιρέσει δύο κάρτες. Εντάξει, τώρα ναι. Εντάξει, σαφές το αποτέλεσμα ότι εγκρίνεται. 54 τώρα παρακαλώ, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία αριθμών 1 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προχωρούμε στην 58, σε τμήματα τώρα. Πρώτο τμήμα για την ψηφοφορία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο, υπέρ. Κατά αποχές επαληθεύουμε το δεύτερο τμήμα. Πέρας της απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές Ας επαληθεύσουμε και αυτό. Την 60 δηλαδή. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ τώρα παρακαλώ. Εντάξει. Πέρα της ψηφορίες. Εγκρίνεται. 59 τώρα. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίν... Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Οι άλλες έχουν καταπέσει. Πάμε στην 63. 63. κατά αποχές επαληθεύουμε. Πέρασε ψηφοφορίες. Εγκρίνονται 64 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η πέντε της αλίας τώρα, σε τμήματα, πρώτο τμήμα. Ευχαριστώ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σε τμήματα τώρα ε, η 11 υπέρ, κατά αποχές, το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12 της ΠΕΣ περ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το, η 8 των αναφορών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 13 της αλίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ενοποιημένη τροπολογία περιθμών 3 τώρα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 11 των αναφορών. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 μπελιέ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και προχωρώ με την 76 και λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επαληθεύουμε την 67. Την 76, συγγνώμη. 76. Πέρα στις ψηφοφορίες. Μάλιστα, απορρίπτεται. Τότε πάμε στην 75 Φανμπρέμπτ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 17 παράγραφος 79 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 των αφορών το τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 80 Κάντμπαχ και λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές επαληθεύμα. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται και πάμε στην 82 και την 83 υπέρ Είναι ταυτόσιμε γι' αυτό, τις ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 85 παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές επαληθεύουμε. Πέρα στις ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Υπάρχει μια παράκληση να ψηφίσουμε την 21 της Αλίας. Έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα. Από τους πράσινους, την κυρία Πελή. Περισμόν 21 της Επιτροπής Αλίας. Δεν νομίζω ότι αυτή η που καλύτερη τροπολογία υπάρχει. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε. Όχι. Λέει η συγγήτρια. Είναι κάτι το οποίο αντιφάσκει σε αυτά τα οποία ψηφίσαμε, λέει η συγγήτρια. Λέει για εθνικούς και τομιακούς στόχους. Θέλουμε μια τέτοια προσέγγιση ένταξη της πολιτικής mainstream και έχουμε τις τροπολογίες από την Επιτροπή Ελίας, την Επιτροπή Αναφορών, γιατί είπαμε ότι θα πρέπει να αφορούν τέτοια θέματα οι επιτροπές της, ε, κάθε επιτροπής, να ασχολούνται με τις τροπολογίες με τις τροπολογίες τις δικές γιατί τα γενικά θέματα, τα γενικά, εμείς τα διεκπεραιώνουμε. Και αυτό και είπαμε, ότι θέλουμε μια ολοκληρωμένη, ολοκληρωμένη προσέγγιση με στόχο το mainstreaming. Και γι' αυτό δεν θέλουμε να έχουμε στόχους ε, σε κουτάκια, εθνικούς στόχους, τομιακούς στόχους. Αργότερα, ναι, θα ζητήσουμε να υπάρχει περισσότερη διασυνοριακή ή τέλο πάντων ευρύτερη συνεργασία. Αν ε, δούμε αυτέ τι τροπολογίε, αντιφάσουν σε όλα όσα κάναμε για άρα να τι αφήσουμε. Ακούσαμε λοιπόν δύο τοποθετήσεις, μία υπέρ και μία κατά τη ψηφοφορία. Τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε εάν θα ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν, παρακαλώ, υπέρ του, να γίνει ψηφοφορία για την 21 η Αλία. Κατά. Αποχές. Μάλλον έχει απορριφθεί. Οπότε φαίνεται το έχει απορρίψει η πλειοψηφία και του δεν γίνεται ε, ψηφοφορία και πάμε στην 87 τροπολογία. πίπτη, μάλλον 89 κατά αποχές απορρίπτεται. Ενοποιημένη τροπολογία υπαριθμών 4. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνεται. Στην 90 τώρα. Όχι, πιο πριν. Πάμε στην 93, δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 93, δεύτερο τμήμα. Πέρα τη πληροφορία. Απορρίπτεται. Με μία ψηφοδιαφορά απορρίπτεται. Στην 90 παρακαλώ, Φαν Μπρέμπτ, με προφορική τροπολογία υπέρ. Η συγκίτρια μια και τη διαβάσαμε το κείμενο, φαίνεται ότι συμφωνεί πολύ καλά, χρήσιμο και αυτό. Υπέρ, κατά λοιπόν τώρα. Αποχές εγκρίνεται. Ενενήντα έξι τώρα, Περέγιο Ροδρίγες, υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 97 Χάμα Πρώτο τμήμα τώρα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 98 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 99 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε το δεύτερο τμήμα. Πέρας τις ψηφορία εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση για το τρίτο τμήμα. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται και περνούμε τώρα σε μια ενοποιημένη τροπολογία, την υπαριθμών 6, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 29 υπέρ, 24 ψήφι κατά. Και έτσι περνάμε μερικές ε, τροπολογίες τα γρήγορα και πάμε στην 88, Γκερμπράντι και λοιπή, υπέρ. Κατά. Αποχές, απόρριπτα. 176, κλάς, υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 27 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 106 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Επαληθεύουμε την 108. Πέρα στις ψηφοφορίες απορρίπτεται. 109 σε τμήματα, πρώτο τμήμα παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 111 με επαλήθευση. Α, επαλήθευση θέλετε. Μάλιστα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Εκατόν έντεκα τώρα υπέρ. Αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Όχι, ήταν σαφές το αποτέλεσμα. 6 της αλίας τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 της αλίας, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 της αλίας, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 119 και 17 της αλίας ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται, 115 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ. 115 λέτε. Όχι, 116 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110, 178 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτωση. Επαλήθευση στην 118. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ηγίτσες. Ε, τέσσερα της Αλίας, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Άποχες. Επαληθεύουμε. Πέρα στις ψηφορίες. Απορρίπτεται. Εκατόν είκοσι εννέα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη τροπολογία υπαριθμών 5 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπότιτλος 6, τροπολογία 130, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. δύο της αλίας υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. δέκα της αλίας υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε τη δέκα της αλίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ταυτόσημες 133-134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 19 της Ελίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. 140 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκατόν σαράντα πρώτο τμήμα επαληθεύουμε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Άρα καταβίπτει και το δεύτερο τμήμα γιατί τελείως δεν έχει νόημα. Και πάμε στην 141 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 144 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απο... Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε το δεύτερο τμήμα. Πέρα τη προφορίες. Εγκρίνεται. 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 158, 160 ταυτόσιμες μαζί υπέρ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Πολυθεύμα. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 162 Φερέιρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 των αναφορών υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 σε τρία τμήματα το πρώτο παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεν ξέρω αν έχει νόημα τώρα να ψήσουμε και το τρίτο. Ναι, το ψηφίζουμε. Τρία, τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 168 απερίφθη, αλλά σε τρία τμήματα. Τρία τμήματα και τρεις φορές ψηφοφορία και να απορριφθεί. Πολύ ωραία. 172 υπέρ, Ε, υπέρ ακόμα. Υπέρ. Ας ξαναρχίσω μπερδευτικά. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται, αλλά να επαληθεύσουμε αν το επιθυμείτε. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚΑ. Πέρασε. Απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 των αναφορών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 189 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 της Ελίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ας επαληθεύσουμε την 20 της Ελίας. Πέρασε ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ. Καταπίπτει 190. Την ψηφίσαμε κιόλας. Καλά. Τότε 191. πράγματι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 της ε, Επιτροπής των Αναφορών δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σκέψει σκέψη μόνο 9 γκροστέτ, τροπολογία γκροστέτ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 αρσένης και λοιπόν, αρσένη και λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές μάλλον εγκρίνεται να το επαληθεύσουμε όμως, το δεύτερο τμήμα. πέρα της φορείες Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Ε, η 12, η Γέκλερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 Ρώση υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 Άντερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 Αρσένης και λοιπόν και λοιποί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπαριθμόν 1 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 16 η, σε δύο τμήματα παρακαλώ πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Επαληθεύουμε το δεύτερο τμήμα. Πέρας προφορίας εγκρίνεται η 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τα καταφέραμε, συγχαρητήρια. Στο σύνολο του ψηφίσματος τώρα η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πω πω, συγχαρητήρια, κοιτάξτε εδώ. 55 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, καμία αποχή και συγχαρητήρια στην Εστέρ Ντελάγκε. Πάει πολύ ισχυρό και καλά προετοιμασμένο το Κοινοβούλιο. Για την COP10 λέει ο Πρόεδρος στην Αγκόγια. Παραμένουμε στη βιοπικιλότητα, στο επόμενο θέμα. Στο 9. στρατηγική στόχη για, το, για τη δέκατη. Συνεδρία έσκεψη των μερών της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα. Υπάρχει προφορική ερώτηση. Την έχετε λάβει. Θα γίνει και συζήτηση στην Ολομέλεια βάσει αυτές τις ερώτησης. Παρατηρήσεις υπάρχουν. Είναι μια πολύ απλή ερώτηση. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Μία φράση είναι όλοι όλοι. Πώς ε, βλέπετε την επίτευξη της επιτυχούς διοργάνωσης της ε, συνέδου αυτής στην Αγκόγια. Άρα εγκρίνεται στο 10 τώρα. Διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων επιπτώσεων. Ja, ich war etwas zu schnell, weil Μάλλον βιάστηκα, λέει ο πρόεδρο. Συνιόριε, σινιόρε. Με ακούει κανείς. Το Ιταλικό, η Ιταλική πτέρυγα του ΕΛΚ ε, έχει αποδειχθεί σε εντατικές συνομιλίες από ό,τι φαίνεται. Yeah. Λοιπόν, εγκρίναμε την ε, ερώτηση μεν, έχουμε όμω και το ψήφισμα. Έχετε το ψήφισμα στο φακελό σα. και ρωτώ ποιος θέλει να λάβει το λόγο για το ψήφισμα. Ουδής. Πολύ καλά. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Άρα θα πει ότι συμφωνείτε όλοι. Το ψήφισμα έτσι για την COP10. Έχουν ζητήσει το λόγο. Μάλλον είναι συντάκτης του ψηφίσματος Σιντελάνγκε, και Κερμπράντι, Μπελιέ, Ουσκί, Λιωτά, Χρόσμπαχ. Κάποιος από τους συντάκτες. Α, η κυρία Μπελιέ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ θετική η δουλειά στο ψήφισμα αυτό. Ξανατονίζω την ανάγκη να έχουμε φιλόδοξη θέση ως Ευρωκοινοβούλιο στην Διεθνή Συνεδρίαση, διάσκεψη μάλλον της Ναγκόγια. Θα ήθελα να επισημάνω τρία σημεία που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο τροπολόγησης και που σας τα προτείνω. Θα ήθελα, εξ ονόματος τη ομάδα των οικολόγων, να επιστήσουμε την προσοχή όσο και αν φαίνεται περίπλοκο διπλωματικά, αλλά είναι σημαντικό, την προσοχή και να καταγγείλουμε την θέση της φιλοξενούσας χώρας στη διεθνή αυτή διάσκεψη για τη βιοποικιλότητα, ενώ την Ιαπωνία και την θέση της όσον αφορά την αλληλεία και την προστασία ορισμένων θαλασσίων ειδών που απειλούνται όπως ο κόκκινος τόνος και η φάλαινα. Συμβολικά και πολιτικά θα πρέπει το Ευρωκοινοβούλιο να εκφράσει την πικρία του και να επιστήσει την προσοχή της Ιαπωνίας να αλλάξει θέση όσον αφορά την αλληλεία. Επίσης, θα θέλαμε σαφώς να αναφερθεί το ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι αντίθετο με την γενίκευση απόλυτα του να δίνονται διπλώματα ευρεσιτεχνίας όσον αφορά τα έμβια όντα. Και η αρχή της αντίθεσης στα διπλώματα αυτά ευρεσιτεχνίας για τα έμβια όντα να αναφέρεται ιδιαίτερα σε σχέση με τις εργασίες που γίνονται για το πώς ε, επιμερίζονται διάφορα πλεονεκτήματα. Και τέλος ένα τρίτο σημείο, τα βιοκαύσιμα. είναι ανάγκη να υπάρξουν κριτήρια δεσμευτικά και βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα. Για αυτά τα τρία σημεία σας καλώ να προσέξετε και επαναλαμβάνω είναι θετικό θετική αυτή η πρώτη δουλειά αυτό το ψήφισμα που ελπίζω να περάσει με πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε τη Σαντρίν Κρήτων. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στα αγγλικά, ο κύριο Αρσένη Συγχαίρω του συντάκτε του ψηφίσματο και θα ήθελα να τονίσω τα εξή. Με βάση τα πρακτικά των δύο τελευταίων συνοδηράσεων μας, ήταν στο Κάλι, Κολομβία, Μάρτιο του 2010, η Βραζιλία και πολλές άλλες χώρες έχουν δηλώσει ότι ενώ το στρατηγικό πρόγραμμα δεν συμφωνούν με ένα στρατηγικό πρόγραμμα 2010-2020 αν δεν υπάρχει σαφής δέσμευση για τη χρηματοδότηση και πρόοδος για την πρόσβαση στο πρωτόκολλο για τα πλεονεκτήματα και ωφέλη μπορούμε να ενισχύσουμε αυτά τα δύο σημεία, νομίζω. Γιατί όπως και στην Κοπενχάγη μπορούμε να διηγηθούμε σε αδίέξοδο στις διαπραγματεύσεις αυτές. Και διάβασα τα πρακτικά και είδα ότι η θέση των ΗΠΑ είναι εσχρή. Και μάλιστα και η θέση της Ένωσης μπορεί να είναι σε αντίθεση με το σημείο 3 της συνθήκης για την δίκαιη κατανομή των του ωφέλους και δεν σέβεται τα δικαιώματα των ε, ηθαγενών και συνθήκη που υπάρχει. Την πρόσβαση και τα δικαιώματα που έχουν για τους ε, ε, ε, ε πόρους, πρόσβαση σε γενετικούς πόρους. Επίσης η Ένωση δεν καλύπτει στην μοίρασμα των γνώσεων. Δηλαδή ουσιαστικά πάμε να αποδυναμώσουμε τις διατάξεις της παρακολούθησης, εντοπισμού και χρήσης των γενετικών πόρων. Το ίδιο και τις... για τη συμφωνία αμοιβαίας χρήσης μεταξύ χρηστών και πάμε. Άλλα λόγια δηλαδή η Ένωση έχει μια θέση που είναι αντίθετη με τις θέσεις των ομάδων εργασίας. Θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για συμφωνία με τους παραδοσιακούς χρήστες των πόρων. Ταυτόχρονα, ως Ένωση, θα έπρεπε να πούμε ότι το πρωτόκολλο αυτό πρέπει να εφαρμοστεί από τη στιγμή που θα επικυρωθεί κι όλοι οι όροι του δεν θα πρέπει να αφαιρέσει κάτι από αυτούς που, έχουν, που είχαν πρόσβαση παραδοσιακά. Επαναλαμβάνω, η θέση της Ένωσης είναι σε εντελώς άλλο μήκος κύματος. Τέλος, κακός έχουμε το CBD ήδη από το 92 Έχουμε δύο άλλες συμβάσεις εμπορικού χαρακτήρα, το ένα για τα φυτικά και γεννητικούς οργανισμούς. Αυτοί κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτοί αναφέρονται στην αγορά, έχουν σχέση με την αγορά. Συνοψίζω, το ψήφισμά μας θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην προσπάθειά μας να πετύχουμε τους στόχους οι οποίοι έχουν οριστεί. Βιτόριο Πρόντι. Δεν θέλει να μιλήσει. Χριστίνα Γκυτάρης Κορτίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το θέμα αυτό για τη βιοποικιλότητα και για το ψήφισμα ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας στη συνάντηση εκείνη που έγινε στη Βόνη. Πρώτα πρώτα, διαπιστώνω στο κείμενο που ψηφίστηκε κάποιες αντιφάσεις. Η μεγάλη μου έκπληξη στη Βόνη ήταν το πρόβλημα των Ιθαγενών και εκείνων που επί τόσο καιρό, επί τόσοι αιώνες, ζουν σε αυτές τις χώρες και τους διώχνουν. Είναι Ινδία, Καμερούν, Αφρική, Μεξικό. Δεν τους αφήνουν να καλλιεργήσουν αυτό το, το, το έδαφος που τους ανήκε ε, ανέκαθεν. Δεν τους αφήνουν να πάνε στους τόπους λατρείας τους τους αρχαίους. Ε, αυτό ήταν κάτι με καταράκωσε. Και βλέπουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πρωτόκολλο και να αναγκάζει σε αντίστοιχη συμπεριφορά αυτούς που έχουν την κυριότητα αυτών των χώρων. Δεν είναι δυνατόν να έχουν τέτοια μεταχείριση άνθρωποι. Πρόκειται για κάποιους που ε, Έχουν κάποιες, κάποιες μεθόδους παραδοσιακές και δεν τους αναγνωρίζουν κανένα, κανένα δικαίωμα. Γι' αυτό στην Ευρώπη αν έχουμε έναν αγρότη που έχει κάποια γη ε, το έχουμε αντίστοιχη συμπεριφορά. Να μην θεωρείτε ότι είναι αμάρτημα η κυριότητα, η ιδιοκτησία της γης. Και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι θα πρέπει να κάτσουμε και να δούμε πώς θα είμαστε συνεπείς. Ότι δηλαδή θα πρέπει οποιοδήποτε χώρος να φροντίζεται. Ε, και ξέρετε με την νομοθεσία δεν γίνεται τίποτα. Θα πρέπει να πιστεί ο κόσμος σύμφωνα με το άρθρο 6 εκείνης της ε, οδηγίας, της οδηγίε Habitat. Και επίσης θα πρέπει κάτι να γίνει με τους αγενείς και θέλω να ζητήσω από την Κομισιόν να βοηθήσει. Είχαμε συναντήσεις με αυτούς τους αγενείς, με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Θα πρέπει να υπάρξει μια τροπολογία και εκεί να απαιτούμε τα παγκόσμια πρωτοκόλλα και του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, αφορούν αυτούς τους χώρους θα πρέπει να συνοδεύονται από την αναγνώριση αυτών των ηθαγενών και των παραδοσιακών τους ε, τρόπων καλλιέργειας της γης. Πρόεδρος, πού ακριβώς διαπιστώνεται ότι υπάρχει αντίφαση στην έκθεση. θα σας τα πω εγγράφως σε, σε ένα κείμενο που θα καταθέσω. Κύριε Κάντμπαχ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Σήμερα με φυσικά όλες τις παρατηρήσεις, παρακαλώ. Μόνο μην ξεχνάτε ότι 15 του μηνός είναι η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών. Βεβαίως, καλό θα είναι να ε, συμμετάσχουν όλοι στην εκπόνηση του εγγράφου, αλλά από την άλλη πρέπει να έχουμε και ένα σαφές κείμενο, να μην χαθούμε σε πολλές λεπτομέρειες και γι' αυτό η προσπάθειά μας θα είναι οι βασικές ιδέες και οι βασικές απόψεις να ενταχθούν ό,τι γράψετε μέσα τροπολογίε θα προσπαθήσουμε να το εντάξουμε στο κείμενό μας χωρίς όμως και να διωγγώσουμε ιδιαίτερα το κείμενο με ιδιαιτερότητε περιφερειακές, τοπικές Και γι' αυτό θα σα παρακαλέσω και αντίστοιχα με τη σημερινή ψηφοφορία για τη βιοπικιλότητα, γιατί ευχαριστώ πολύ επί τη ευκαιρία για την ε, στάση σας στις ψηφοφορίες, είναι καλό να μην ε, νερώνουμε υπερβολικά τα κείμενά μας, να έχουμε πιο επικεντρωμένη παρουσία των θέσεών μας. Πρόκειται για ψηφίσματα ε, τα οποία εκθέτουν στον έξω κόσμο τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βεβαίως πρέπει πάντα να καταγράφουμε τα ουσιοδέστατα συμφέροντα των ομάδων των εμπλεκομένων πληθυσμών ή ηθαγενών και γι' αυτό καλό θα είναι πάντοτε να ενισχύουμε αυτή τη διάσταση και ταυτόχρονα πρέπει να κερδίσουμε και τους πολίτες. Ε, πράγμα το οποίο ακόμη ίσως δεν έχουμε εξασφαλίσει, δηλαδή δεν ε, υπάρχει η διάθεση να ενσωματωθεί η προστασία των ειδών, η βιοπικιλότητα σε όλα στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως θα έπρεπε. Η διαφύλαξη της βιοπικιλότητας, η προστασία των ειδών δεν φαίνεται να έχει εγγραφεί σε κάποιο είδος πολιτικής ώστε να έχουμε απτά αποτελέσματα χωρίς και πολλές δαπάνες σε τελευταία ανάλυση. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική μας τάση ε, στο ψήφισμα αυτό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και την γραμματεία για το ψήφισμα αυτό με την Αγκόλια. που έγινε και με ανταλλαγή email κλπ. Έγινε λοιπόν με μεγάλη ταχύτητα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και συμφωνώ και με τη συνάδελφο Κάλεμπαχ. Θα πρέπει να φροντίσουμε το θέμα αυτό και το ψήφισμα αυτό να μην υπερδιαβρυνθεί. και τελικά να πνιγεί η φωνή μας. Πρέπει να εκφραστούμε με μία φωνή, είναι σημαντικό αυτό. Τώρα, οι προτινόμενες προσθήκες, η, δηλαδή, η ανθρώπινη διάσταση του συναδέλφου ΕΛΚ, αλλά και της Αντρίν Μπελιέ για την αλληλεία του τόνου, του κόκκινου τόνου και της φάλαινας. Όντως, έχουμε δώσει μάχες στο Ευρωκοινοβούλιο γι' αυτό και πρέπει λοιπόν τα σημεία αυτά να μπουν στο ψήφισμα και να υποθούν στην Ιαπωνία, προς την Ιαπωνία. Τώρα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τα έμβια Είναι σημαντικό οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την διαφορότητα η οποία υπάρχει και να μην περάσουν τα δικαιώματα αυτά και τα ωφέλη στις πολυεθνικές. Πρέπει να βρούμε τον σωστό τρόπο διατύπωσης. Αλλά το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε προς την Κομισιόν είναι πώς η Κομισιόν θα φροντίσει να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη που κάναμε στις μεγάλες διεθνείς διασκέψεις και να μην τρώμε ώρες και ώρες και ώρες να συζητάμε μεταξύ μας ενώ οι άλλες χώρες έχουν συμφωνήσει στα, στα περιθώρια της διάσκεψης μεταξύ τους. Το πιο σημαντικό επαναλαμβάνει το μήνυμα που θα πρέπει να στείλουμε προς την Ιαπωνία. Καλώς, θα ήθελα να ρωτήσουμε κατευθείαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα τα καταφέρετε να μην είναι μόνο για το Θεαθήνα η εμφάνισή σας, αλλά να έχετε ουσιαστική παρουσία κύριος Κρός είναι εδώ. Να δούμε τι έχει να μας πει. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την προετοιμασία. Δύο λόγια τι γίνεται με τον εσωτερικό συντονισμό που μόλις τώρα ξεκίνησε με τη Βελγική Προεδρία. Είχαμε ήδη μερικές συναντήσεις και στο Κάλι και στο Ναϊρόμπι. Με βάση όλα αυτά έχουμε την εσωτερική διαβούλευση τώρα και με όλα τα κράτη-μέλη. Προετοιμάζουμε τη θέση της Ένωσης. Έχουμε ειδικέ επαφές με τη Βελγική Προεδρία. Είχαμε και θα οριστικοποιήσουμε τη θέση αυτή για τα πορίσματα του Συμβουλίου τον Οκτώβριο, γύρω στα μέσα Οκτωβρίου. Και θα ενημερώσουμε και τους βουλευτές για τις προετοιμασίες αυτές λίγο αργότερα. Ενδεχομένως στις αρχές Οκτωβρίου να συναντηθούμε να σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το που θα βρισκόμαστε τότε. Τώρα για το μοίρασμα πρόσβασης και ο ωφέλους, οι τελικές διαπραγματεύσεις γίνονται αυτή τη βδομάδα στο Μοντρεάλ. Θα πρέπει να περιμένουμε και αυτά τα αποτελέσματα από εκεί, γιατί είναι ένα πακέτο θεμάτων που θα συζητηθούν στην δέκατη συνάντηση στην Αγκόγια. Με το στρατηγικό στοχο στόχος βιοποικιλότητας 2010-2020, επιμερισμός των εκτιμάτων και πρόσβασης και φυσικά η χρηματοδότηση. Το ελμίζω θέμα και αυτό. Αυτή τη βδομάδα έχουμε παραλαμβάνει τη συνάντηση στο Μοντριάλ και με βάση τα πορίσματα αυτά θα ξαναδούμε το πακέτο. Πρόεδρος, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση προς την Κομισιόν. Ξέρω και καταλαβαίνω ότι χρειάζεται χρόνος να πετύχουμε κοινή θέση ω Ένωση. Λέτε θα υπάρξει κοινή θέση μέσα Οκτωβρίου. Ξέρουμε ότι τέλος Οκτωβρίου είναι αγκόγια. Πολύ φοβάμαι ότι θα κάνουμε το ίδιο λάθος που κάναμε και στην Κοπεχάγη και στην Τόχα κλπ. Δηλαδή η συγκεκριμένη μου ερώτηση είναι τι κάνουμε τώρα, τώρα. Σε σχέση με άλλες χώρες εκτός Ένωσης και οι χώρες αυτές να συμπλέψουν με μας. Ή και πάλι θα περιμένουμε να έχουμε την κοινή θέση μέσα Οκτωβρίου, θα πάμε στην Αγκόγια και να δούμε ότι όλες οι άλλες χώρες ήδη έχουν άλλη θέση. Τι κάνουμε τώρα για να φέρουμε και άλλες χώρες στη δική μας ρότα. Ευχαριστώ. Κρήτον Αρσένης, μια ερώτηση. Δεν θα μοιάζει με την Κοπεχάγη ιδιαίτερα όσον αφορά στην πρόσβαση και στο επιμερισμό των δικαιωμάτων, αν δεν το πετύχουμε να φέρουμε και άλλες χώρες κοντά μας, θα είναι χειρότερα. Και θα ήθελα η Κομισιόν να επιβεβαιώσει αυτά που είπα, αληθεύουν, για τις επιφυλάξεις που έχει η Κομισιόν στο να αναφερθούν τα δικαιώματα και η ιδιοκτησία των πιθαγενών κοινοτήτων, πόρους να μην υπάρχει προειδοποίηση εκ των προτέρων και προσπαθεί να αποδυναμώσει το μηχανισμό εθελοντικής χρήσης, συμφωνία για τις αμοιβαία αποδεκτές συμφωνίες. Το είπα και πριν και θα ήθελα παρακαλώ η Κομισιόν να το σχολιάσει αυτό. Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα για το τι κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτές τις τρίτες χώρες. Λίγο πριν την κόπη διαμορφώθηκε η κοινή θέση, αλλά τώρα που μιλάμε, έχουμε μια συνάντηση στο Μόντρελ για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τους εμπλεκόμενους και να δούμε πού μπορούμε να κλείσουμε κάποιους συμβιβασμούς επί τη βάση των θέσεων που είχαμε διαμορφώσει. Επομένως, βλέπετε, ότι έχουμε αυτές τις άτυπες επαφές που γίνονται στα περιθώρια των συναντήσεων. Όπως έγινε και τον Απρίλιο, προσπαθούμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να εξηγήσουμε τις θέσεις μας στους συνομιλητές μας. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε την συνάντηση ψηλού επίπεδου του Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη Ε, θα γίνει αυτή η συνάντηση στον ΟΗΕ για την βιοποικιλότητα. Θα παραστούν ε, υπουργοί, θα υπάρξει προετοιμασία για την ε, ΚΟΠ στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Και σε εκείνη τη συνάντηση θα είναι και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ελπίζουμε να επιδευτεί συμφωνία στα βασικότερα ζητήματα και επομένως και πριν την κόπη κάποια θέματα να έχουν επιληφθεί τρόσον αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αυτό το οποίο αναφέρθηκε Σας είπα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στο Μόντριελ δεν έχω ενημερωθεί ακόμα. Δεν μπορώ να σας πω τι συζητείτε τώρα στο Μόντριελ πώς διαμορφώνονται οι θέσεις και πού πάει το πράγμα για τους ηθαγενείς τώρα και τα δικαιώματά τους και όσον αφορά τι προδοσιακές μορφές γνώσεις θα πρέπει παραδοσιακή γνώση να αναφερθεί στο πρωτόκολλο για αυτούς τους ηθαγενείς τις τοπικές κοινότητες επίσης αυτό το οποίο προωθούμε είναι κάποιες διατάξεις για να δεσμεύονται οι χώρες για κάποιους μηχανισμούς που θα επιτρέψουν στους Ιθαγενείς ε, να εμπλακούν στις διαπραγματεύσεις. Αυτό βέβαια θα αφορά την εθνική νομοθεσία ή θέσπιση τέτοιες υποχρέωση. Γίνεται πολιτική ζήμωση πάνω σε αυτό. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει κάποιες θέσεις και άλλοι ενδιαφέρονται. για το τι θα γίνει στο πρωτόκολλο. Και όσον αφορά αυτές τις υποεξέλιξη διαπραγματεύσεις, το συντομότερο δυνατόν θα σας ενημερώσουμε ακριβώς όπως έγινε και στο παρελθόν. Πριν από λίγες εβδομάδες. Δυστυχώ δεν είναι εδώ οι αρμόδιοι συνάδελφοι να σα πούν περισσότερε λεπτομέρειε. Ευχαριστώ, δεν στέκει κανεί άλλο το λόγο. Ευχαριστώ του συντάκτε του ψηφίσματο λοιπόν. Και όπω είπαμε, προθεσμία για την καταστροφή λογιών αύριο στι 10. Και θα πρέπει να είναι σχετικά σύντομο το ψήφισμα όπως ακούσαμε. Τελευταίο σημείο για σήμερα το πρωί. Ναι, και το 11 το Είδαμε ήδη το, την αποκεντρωμένη υπηρεσία της ΕΦΣΑ δηλαδή. Έχουμε τώρα το 10 της ανεξάρτητων εκτιμήσεων επιπτώσεων. Ο κύριος Κάλαραν είναι ο συντάκτης γνωμοδότηση για την Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων. Ο κ. Χάλλαν, παρακαλώ. Not the, uh, uh, most... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως σωστά είπες Πρόεδρε, έχουμε αυτή τη γνωμοδότηση προς την Επιτροπή ε, Νομικών Θεμάτων για τη διασφάλιση ανεξαρτήτων εκτιμήσεων επιπτώσεων και η κυρία Νίμπλερ έχει αναλάβει την γνωμοδότηση για την νομική επιτροπή. Και συμφωνώ με κάτι το οποίο αναφέρει στο τελικό του, δηλαδή η Κομισιόν θα πρέπει να φέρει την τελική ευθύνη για αυτές τις ε, εκτιμήσεις επιπτώσεων, αλλά θα πρέπει να περνάνε από έλεγχο ποιότητας. Άρα να εκμεταλλευτούμε την πείρα, τη γνώση της ε, Επιτροπής. Όμως θα πρέπει επιπλέον να υπάρχει ανεξάρτητος, αμερόληπτος, εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος και αυτό θα γίνει αν συγκροτηθεί μια επιτροπή που θα κάνει αυτή τη δουλειά για τις ε, εκτιμήσει εκτιμήσεις της Επιτροπής. Ε, Η Βασίλειο κάτω χώρε, Γερμανία, Σουηδία έχουν τέτοιες επιτροπές που κάνουν αυτή τη δουλειά. Έχω λάβει από διάφορους εμπλεκομένου ε, διάφορα σχόλια. Υπάρχει προβληματισμό θεμητό κατά τη γνώμη του όσον αφορά αυτές τι εκτιμήσεις τη επιτροπή, που πολλές φορές είναι κομμένες και αραμένες για κάποια απόφαση που ήδη έχει ληφθεί και δεν γίνονται αυτέ οι εκθέσει αυτέ οι εκτιμήσει για να βοηθηθεί η λήψη απόφαση. Επίσης, θα ήταν σωστό η Επιτροπή μας να κάνει ό,τι κάνει η κυρία αρμόδια ΙΜΚΟ. Με το που αρχίζουν οι ανταλλαγές ε, με την Επιτροπή για κάποια πρόταση. Και να κάνουμε για εμείς την αξιολόγησή μας για τις τυχόν αν θέλουμε να κάνουμε τροποποίηση και με τις τροπολογίες τότε θα πρέπει και εμείς να έχουμε το θάρρος να προβαίνουμε σε τέτοιου είδους Γιατί πολλές φορές πρόκειται για κάποια ουσιώδη ζητήματα. Και επομένως, πριν εγκρίνουμε κάτι, να μπορούμε να έχουμε κάνει αξιολόγησή μας, γιατί νομίζω ότι είναι πιο σωστό να υπάρχει ευρύτερη ε, ζήμωση με τους ε, ε, εμπλεκόμενους, να έχουμε κάποια ανάλυση κόστος ωφέλους. Και να κάνουμε κάτι όταν χρειάζεται. Πολλές φορές θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δύσκολο μετρήσιμες και επιπτώσεις. δεν μετρούνται όλα με, νούμερα και με κόστος και το κόστος και το όφελος τα οποία ε, κόστος και όφελος θα πρέπει να ε, εξηγούνται καλά. Νομίζω επομένω ότι οι εκτιμήσει για ανεξάρτητε είναι πάρα πολύ βασικέ και μπορούν να διαμορφώσουν τη θέση μας όσον αφορά την νομοθεσία, αλλά το κλειδί για όλα αυτά είναι ότι θα πρέπει να είναι ανεξάρτητε αυτέ οι εκτιμήσει το κλειδί για την επιτυχία του εγχειρήματος. Ευχαριστούμε κύριε Καλά. Άρα, σε τέτοια περίπλοκα ζητήματα, καλό θέλει να έχουμε μια ιδέα των επιπτώσεων. Αξιολόγηση επιπτώσεων λοιπόν πρέπει να υπάρχει. Έχουμε την εντύπωση όμως ότι μερικές φορές αυτή γίνεται με τρόπο που να δικαιολογεί την ύπαρξη των εγγράφων περισσότερο. Λίγο πολύ. Δηλαδή, να εξυπηρετηθεί η σκοπιμότητα του συντάκτη ενός ομοθετημάτους. πράγμα το οποίο δεν είναι το σωστό. Έχουμε πει ότι σε περίπτωση τροποποίηση νομοθεσία πρέπει να γίνεται με την Επιτροπή και το Συμβούλιο ε, η αξιολόγηση των επιπτώσεων του νομοθετήματο. Εμεί, όπω βλέπετε, είμαστε κάπω διστακτικοί ω προ την εκτίμηση των συνεπειών ως νομοθέτες του άλλους έχουμε την δυνατότητα, έχουμε την ελευθερία να αποκλίνουμε από την αξιολόγηση αυτή, όσο και αν διστάζουμε μερικές φορές να το κάνουμε την ώρα της αλήθειας. Παρακαλώ, κυρία Κουτιέρης Κορτίνας. Eh, έχουν φύγει προς συνάδελφοι, αλλά με εκπλήσει το ότι το σημείο κλειδί είναι αυτή η αξιολόγηση. Επίπτωση είναι η λέξη κλειδί. Επίπτωση σε σχέση με την νομοθεσία της ε, Ένωσης. Να, τι διάκριση πρέπει να γίνει. Αυτό που είπε η κυρία Νίμπλερ. Πολύ δημοκρατικό αυτό. Δεν, δεν επιβάλλει τίποτα. Ερωτά, προβληματίζεται. Επομένως, γενικά για ε, απασχόληση, οικονομία κλπ. Ποια είναι η επίπτωση των όσων κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο κάνει την ε, αξιολόγηση, τι συμφέροντα έχει, με τι κριτήρια γίνεται αυτό. Να είναι τρει ερωτήσει που θα μετρήσουν τα επόμενα χρόνια γιατί ε, του χρόνου πρόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να κάνει την αναθεώρηση της οδηγίας για το περιβάλλον. Άρα, πρώτον, το θέμα το κανονιστικό. Οι ερευνητικές επιπτώσεις του κοινοτικού δικαίου έχουν φανεί και είναι φυσιολογικό γιατί υπάρχει πολυνομία και πολλές φορές η Κομισιόν κάνει ό,τι θέλει, δεν, δεν, δεν εξετάσει τίποτα εκλογέ. Και επομένως η Κομισιόν δεν, δεν της αρέσει, δεν, δεν σηκώνει κριτική, δεν της αρέσει κριτική. Άρα χρειάζεται να υπάρχει κάποιος ανεξάρτητος που να κάνει αυτή την αξιολόγηση. Μπορεί κανείς να έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι. Να, με το ρίτσι δεν τι έγινε. Άρα να προσέξουμε πώς θα γίνεται η διαδικασία. Θέλω να είναι ανεξάρτητη η αξιολόγηση, όμως κάτι παραπάνω. Εγώ θα έλεγα ότι σε εκείνα, ε, εκείνοι που θα ωφεληθούν σε κάποιες χώρες από μια πρωτοβουλία ε, αυτοί θα πρέπει να κρυθούν από κάποιον εξάρτητο για τις επιπτώσεις. Χωροταξία στην Ισπανία. Η... Τι να σας πω... Ε, έχω, έχουμε αυτό τα, όλα αυτά τα, τα, βουνά από, από, από τσιμέντο τα οποία σηκώνονται ξαφνικά από, τις, ε, από τους εργολάβους και πολλές φορές δεν υπάρχει κάποιος να κάτσει να, να, κάνει τις επιπτώσεις γιατί δεν έχει προϋπολογισμό. Επομένως, τι γίνεται, ποιος ωφελείται, ποιος δίνει τις άδειε ανοικοδόμησης. Πολλές φορές μας ε, κατηγορούν άδικα, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε κανείς να υπάρχει επίκριση. και πολλές φορές υπερβάλλουν όσον αφορά την ενοικοδόμηση κάποιες τοπικές αρχές γιατί έτσι αποσπούν κάποια κονδύλια. Και τελικά ποιος ωφελείται αυτός ο οποίος δίνει τις άδειες ενοικοδόμησης. Γι' αυτό και εγώ σας λέω ότι το σωστό είναι αυτό το οποίο είπε ο φίλος Κάλαναν. Και επιπλέον θα πρέπει ε, να υπάρχει κάποιο είδου αυτοκριτική της Κομισιόν όσον αφορά την νομοθεσία που θεσπίζει. Ε, υπάρχει ένας φορέας νορβηγικός, ανεξάρτητος φορέας, που μπορεί να κάτσει να δει τι γίνεται όσον αφορά την νομοθεσία του περιβάλλοντος της, ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχουν γίνει ένα σωρό απαγορεύσεις που έχουν κάνει πάρα πολύ κακό. Μέταλλα, μόλιβδο. Ε, ε, και αυτό έχει, έχει χτυπήσει πάρα πολύ τη, τον τομέα των εστιατορίων, τον κλάδο των εστιατορίων. Και αυτό είναι υπερβολικό. Και κάθονται α πούμε, και λένε για κάποια μέταλλα που υπάρχουν σε κάποια μουσικά όργανα. Και αυτά θέλουν να τα απαγορεύσουν, αλλά αυτά υπάρχουν από την εποχή του Μπαχ. Επομένω θα πρέπει να κάτσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρήσει και να δει ποιε είναι οι επιπτώσει. Μπορεί να υπάρξουν κάποιε εξαιρέσει που δεν κοστίζουν τίποτα. Να μην είμαστε δογματικοί. Δεν πρόκειται εδώ περί θρησκείας. Άρα και εγώ θέλω πρώτα πρώτα να υπάρχει ε, έκθεση επιπτώσεων πρώτον ανεξάρτητη, δεύτερον θα πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ ακριβής όσον αφορά τις επιπτώσεις όπως ας πούμε για την περίπτωση του περιβάλλοντος και όπως είπαν οι συνάδελφοι, με μια task force να παρακολουθήσουμε το τι γίνεται γιατί είναι κάτι το οποίο αγγίζει την καθημερινή ζωή και είναι κάτι το οποίο αφορά γενικότερα όλη την πολιτική του περιβάλλον. Uh, Ευχαριστώ. Λέει κυρία Πάρα πολύ σημαντικές είναι αυτές οι αξιολογήσεις, ιδίως για την φάση τώρα, μετά δηλαδή τη συνθήκη της Λισαβόνα και εμείς επομένως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την καλή ποιότητα και το ότι να γίνονται από κάποιον ανεξάρτητο. Να σου πω τις θέσεις των σοσιαλιστών πάνω σε αυτό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να κατευθύνουν αυτές οι αξιολογήσεις την νομοθεσία ε, αλλά να μην εμποδίζουν τον ρόλο του νομοθέτη που έχει την πολιτική ευθύνη και να την υπόψη όχι μόνο οικονομική, οικονομικά κριτήρια αλλά και περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικά. Να κάτσουμε και να δούμε ποιες προτάσεις ε, χρειάζονται τέτοιες αξιολογήσεις. Ε, κάποιες φορές τα πράγματα είναι απλά, κάποιες άλλες φορές τα πράγματα είναι περίπλοκα. Άλλοτε δεν πήγουν τα πράγματα, άλλοτε πήγουν πολύ περισσότερο. Εγώ πάντως ε, θεωρώ ότι θα πρέπει αυτό να είναι υποχρεωτικό για κάθε πρόταση. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η άριστη πρακτική, ε, ε, τι επικρατεί στα κράτη-μέλη. Σε Γερμανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε εξωτερικού φορεί, όπω ήδη προαναφέρθηκε για τέτοιε αξιολογήσει. Άρα να κάτσουμε και να δούμε τι μπορούμε να διδαχθούμε από την εμπειρία αυτών των κρατών. Και αυτή η η ανεξάρτητα εκτίμηση θα πρέπει να εξετάζει το, τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων, πώς είναι δυνατόν να αποφύγουμε τη σύγκρουση ε, συμφερόντων. Γιατί πολλές φορές ανακύπτουν τα ζητήματα αφού έχει γίνει η εκτίμηση, αφού έχει γίνει η ζημιά. Σε με την ε, πρόταση ε, ότι από την εκτίμηση θα, εξαρτάται το αν το κοινοβούλιο θα λέει ναι ή όχι σε κάποια νομοθετική πρόταση, δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να μα υποδεικνύει κανεί θέματα. θα, θα αποφασίσουμε. Εμεί είμαστε πολιτικά υπεύθυνοι και εμεί είμαστε αρμόδιοι μόνοι για τι πολιτικέ αποφάσει. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την γνωμοδότηση και του αμέσω επόμενου μήνε ελπίζω θα συνεργαστούν. Σάτουχας. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia raportöörille Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανα. Το καλύτερα. Θέλω και εγώ να υπογραμμίσω ότι η των επιπτώσεων δεν μπορεί να πιέσει προς συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων απλώς βελτιώνει την βάση, την πληροφόρησή μας, τη βάση πάνω στην οποία λαμβάνουμε αποφάσεις. Η ε, συντάκτης της εκθέσεως εκ μέρους της Επιτροπής των Νομικών Υποθέσεων, η κυρία Νίπλερ, έχει υπογραμμίσει τρία σημεία σαν βασικά χαρακτηριστικά αυτής της αξιολόγησης που και πρέπει, εμείς θα πρέπει νομίζω να περιλάβουμε να ακολουθήσουμε στη γνωμοδότησή μας. Η αξιολόγηση λοιπόν είναι καταρχάς ένα μέσον υποστήριξης ε, της πολιτικής αποφάσεως και δεν μπορούν ποτέ να υποκαταστήσουν μια πολιτική απόφαση. Επίσης δεν μπορούν ποτέ να περιορίσουν μια πολιτική απόφαση αυτές οι εκθέσεις αξιολόγησης, οι μελέτες αξιολόγησης, ούτε να παρεμποδίσουν τη λήψη μιας απόφασης. Δηλαδή, ο νομοθέτης διατηρεί την εξουσία και το δικαίωμα, όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε δημοκρατικό καθεστώς. Ο κ. στο σημείο 5 της νομοδότησής του, προτείνει μια υποχρεωτική ανάλυση κόστους και ωφέλους. Με τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα εκπεφρασμένα σε όρους κόστους. Και εδώ διαφοροποιείται από τις θέσεις της κυρίας Νίμπλερ, τις γενικές θέσεις. Και εγώ θα ακολουθήσω την κυρία Νίμπλερ. Υπάρχουν ε, πολλά σημεία στα οποία δεν μπορούμε να ποσοστοποιήσουμε, να προσμετρήσουμε με όρους οικονομικούς το κόστος ή το ε, κέρδος. Αν μιλούμε για ε, υγεία, δημόσια υγεία, περιβάλλον, πώς μετριέται αυτό η ποιότητα της δημόσιας υγείας, πώς μπορεί να μετρηθεί σε οικονομικούς όρους. Και ένα άλλο πρόσφατο παράδειγμα για τις οικονομικές ε, επιπτώσεις που έχουν αξιολογηθεί ε, σε σχέση παραδείγματι με τις επιπτώσεις εναλλακτικών υλικών δεν είναι δυνατόν πάντοτε να προσμετρούνται αυτές ε, οι επιπτώσεις. Εάν, ε, παραδείγματι, θέλουμε να δούμε τι είδους συνέπειες μπορεί να έχει κρίση κάποιου υλικού στην βιοπικιλότητα για τη λαξία ενός είδους. Το ίδιο ισχύει και για, την, ε, για τον άνθρωπο, για, τον, για την ανθρώπινη ζωή. Με τους υπολογισμούς μας είναι δυνατόν, όση αξία υψηλή και να δώσουμε στην ανθρώπινη ζωή, είναι δυνατόν ποτέ να πούμε αξίζει τόσα χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν οι αναλύσεις αυτές αναγκαστικά κάποτε θα γίνονται και αφαίρετες, ε, αναγκαστικά ε, θα, θα στηριχθούν μόνο σε ποσοτικούς αλλά και σε ποιοτικούς ε, δείκτες. Επίσης, εκεί που λέει ο κύριος Κάλαχαν ότι θα πρέπει να συμμετέχουν και οι επιτροπές του, θα πρέπει να λαμβάνουν την απόφαση αν χρειάζεται μια αξιολόγηση οι επιτροπέ του Κοινοβουλίου. Εδώ όμω έρχεται σε αντίθεση ο κ. Κάλλαν με τα όσα προτείνει η κυρία Νίμπλερ στην Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων. Γιατί δείχνει ότι ο νομοθέτης μπορεί να μην διαθέτει όλη την ελευθερία κρίσεως που θα έπρεπε να έχει ένας νομοθέτης σε δημοκρατικό πολίτευμα ο κύριος Κάλλαραν λέει να προσανατολισόμαστε προς την διοργανική συμφωνία, αλλά νομίζω ότι ε, την καθιστά πιο δεσμευτική από ό,τι πραγματικά είναι, γιατί η διοργανική συμφωνία λέει ότι αν τα νομοθετικά, τα αρμόδια για την νομοθεσία όργανα θέλουν να επιφέρουν ε, συγκεκριμένες ε, ε, ριζικές αλλαγές στο νομοθέτημα, τότε μπορεί να γίνει αξιολόγηση επιπτώσεων και δεν, δεν την αναφέρει όμως ως υποχρεωτική, όπως λέει ο κύριος Καλάραν εδώ δυνατότητα δηλαδή προσφέρεται και δεν θέλουμε να περιορίσουμε τις επιλογές μας ως κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε δηλαδή να το καθαταστήσουμε αυτό υποχρεωτικό. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια καλή ισορροπία μεταξύ των επιδιώξεων του κυρίου Κάλαναν για καλύτερες στο βαθμό του δυνατού ε, συνθήκες για τη λήψη των αποφάσεων και του δημοκρατικού πολιτεύματος και τη δυνατότητα να διαφυλαχθούν οι δημοκρατικές συνθήκες ε, για τη λήψη των αποφάσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρόντε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον συνάδελφο Κάλλαναν. Αν και με προβλημάτισε κάπως το θέμα. Η Ένωση έχει εργαλεία στα χέρια της Και πρώτα αυτά πρέπει να χρησιμοποιήσει και ζητήσει να, έχει, να αποκτήσει και άλλα εργαλεία. Εξηγούμε. Η Κομισιόν είναι αρμόδια και μπορεί να χρησιμοποιήσει τα θέματα εμβάθυνση στο κοινό κέντρο έρευνας που εξαρτάται από την Κομισιόν. επαναλαμβάνω για εμβάθυνση θεμάτων. Η Κομισιόν ως εκτελεστικός βραχίωνας και με το δικαίωμα που έχει να προτείνει νομοθετήματα μπορεί να χρησιμοποιήσει το κέντρο αυτό. Αυτό είναι ένα το κρατόμενο. Είναι ένα όργανο το οποίο δουλεύει πολύ εμπεριστατωμένο. Μετά έχει τις υπηρεσίες, διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς. Πιο πριν μιλήσαμε για την ΕΦΣΑ. Στην επίσκεψη που κάναμε, επιμείναμε ιδιαίτερα στην ανεξαρτησία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΦΣΑ. Πριν λοιπόν ζητήσουμε εξωτερική βοήθεια, να αναλύσουμε το σύστημα των οργάνων και υπηρεσιών που έχουμε, να είναι ανεξάρτητες. Παραδείγματος χάρη, ο οργανισμός, η υπηρεσία για το περιβάλλον της Κοπενχάγης έχει υποδομή άκρος επαγγελματική ανεξάρτητη από ό,τι ξέρω. Μπορούμε να έχουμε επαγγελματίες ανεξάρτητους στην υπηρεσία που να επιφορτιστούν με αυτό το έργο αξιολόγησης επιπτώσεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν επαγγελματίες εκτός της Κομισιόν στην Ευρώπη, τουλάχιστον που μπορούν να συγκριθούν με την υπηρεσία για το περιβάλλον της Κοπεχάγης. Άρα πριν ζητήσουμε βοήθεια ή πριν συστήσουμε εξωτερικούς οργανισμούς μας διερωτηθούμε οι υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν και που διαθέτουμε είναι επαρκώς ανεξάρτητες και πρέπει να είναι. Γιατί εμείς ανέκαθεν επιμένουμε στην ανεξαρτησία των διοικητικών συμβουλίων των υπηρεσιών αυτών. Υπάρχει λοιπόν ο άκρος επαγγελματικός χαρακτήρας και εξειδίκευση των υπηρεσιών αυτών. Αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι υπεύθυνε για την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Για συγκεκριμένα κατεξαίρεση θέματα μπορούμε να ζητήσουμε να προσθεθούν και μέλη που θα τη χάνουν της εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι ο κανόνας. Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητάει, να ζητήσει μάλλον, προσωπικότητες που εμεί θα αποφασίσουμε ποιες θα είναι, να εμπλουτίσουν τα διοικητικά συμβούλια ή επιμέρους εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών αυτών. Να δημιουργεί ένα είδος συμβούλιο των υπηρεσιών αυτών, γιατί είναι πολλές αυτές οι υπηρεσίες που ασχολούνται με το περιβάλλον επαναλαμβάνω πρόκειται για πάρα πολλού, πολύ καλούς επαγγελματίες. Και μπορούν να οργανωθούν οι υπηρεσίες αυτές έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο έργο αξιολόγησης επιπτώσεων στο περιβάλλον. Υπάρχουν πάρα πολύ και πλούσιοι ανθρώπινοι πόροι στην Ένωση. Ε, ας τις χρησιμοποιούμε. Και να είναι ανεξάρτητες οι δυνάμεις αυτές. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω τους συναδέλφους οι οποίοι ασχολήθηκαν με αυτό το περίπλοκο θέμα διότι εδώ τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα όσον αφορά το τι θα γίνει με τις εκτιμήσεις επιπτώσεων για την νομοθετική διαδικασία. Εγώ θέλω να σταθώ στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και όσον αφορά τις ε, εκτιμήσεις νομίζω ότι πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τον παράγοντα περιβάλλον. Τα αποτελέσματα στο περιβάλλον για ε, που μάλλον θα, θα, προκύψουν για κάποιο ε, νομοθέτημα ή από κάποιο νομοθέτημα και να ληφθεί υπόψη το τι λέει η, εκτίμηση για το αν θα πούμε το νέο έξι ένα νομοθέτημα και αυτό θα πρέπει να αφορά κάθε οικονομική δραστηριότητα. Ε, επομένως θα πρέπει να δούμε αν, υπάρχει, αν υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Κάποια αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Θεωρώ ότι οι πολίτες της ε, Ένωσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εμείς χρησιμοποιούμε και βασιζόμαστε σε κάποιους ανεξάρτητους και μιλώ τώρα και για την ενεργειακή πολιτική αλλά και για άλλες. Μέχρι σήμερα είναι έτσι η κατάσταση που αναθέτει η Επιτροπή σε κάποιε εταιρείε να κάνουν κάποια ανάλυση, κάποιε εκτιμήσει. Κάποιες φορές όμως αυτές οι εκτιμήσεις συγκαλύπτουν κάποιες παράνομες δραστηριότητε. Γι' αυτό έχει σημασία αυτός που κάνει τις εκτιμήσεις να είναι ανεξάρτητος, να είναι αμερόληπτος σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Άρα ε, θα πρέπει περισσότερο να ασχοληθούμε όσον αφορά την, ε, ε, τις επιπτώσεις της οδηγίας για το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Παρακαλώ την Επιτροπή να λάβει θέση στο θέμα αυτό. Ε, thank you, Mr. Chairman. Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, εμείς έχουμε δεσμευτεί να έχουμε ποιοτικέ εκτιμήσει επιπτώσεων, γι' αυτό και συμφωνούμε με το σχέδιο νομοδότηση. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα απόσπαστο τμήμα τη ε, δουλειά μα και πάντοτε ε, λαμβάνει λάβανε υπόψη όλα όσα είπαν οι βουλευτέ. Το πρόβλημα είναι κατά πόσο κάποιο εξαιρετικό θα συμμετέχει στι εκτιμήσει τη ε, δουλειά μα, που δεν θεωρούμε ότι είναι σωστό. Γιατί διότι θεωρούμε ότι η Επιτροπή Εκτιμήσεων ε, είναι ανεξάρτητη, ε, συμμετέχουν, ε, σε οικονομικ... συμμετέχουν κάποιοι που έχουν ταψαντήσει τις διευθύνσεις και κοιτάνε τις οικονομικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επομένως και άκουσε τι ελέγχθη για το ότι υπάρχουν σε κάποια κρατημέλη ανεξάρτητοι φορείς που όμως τελικά προσανατολίζονται προς ε, τις επιχειρήσεις, άρα αυτό δεν είναι τόσο παράδειγμα προς μίμηση, γιατί εμείς θέλουμε από τα οικονομικά που ασχολούνται περισσότερο αυτές οι εθνικές ε, επιτροπές, να κοιτάμε τα, και τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά. Ο πρόεδρος ορίζει κάποιους να κάνουν τις εκτιμήσεις ε, ανεξάρτητα από τη δουλειά τους της γενικές διευθύνσεις Επομένως πριν εγκρίνει κάποιο κείμενο η Κομισιόν έχουν, έχουν γίνει αυτέ οι εκτιμήσεις. Η εξωτερική όμως είναι δύσκολο να κάνουν αυτή τη δουλειά όπως ας πούμε κάποιοι από το, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε του σωστό να εμπλακούν στην δική μας δουλειά. είναι κάποια πράγματα ιστορικά δικά μας, οπότε πώ θα έρθει κάποιο εξωτερικό να, να τα χτενίσει, να τα ελέγξει. Επίση λέμε ότι θα πρέπει να εξασφαλίζει η Κομισιόν ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων θα πρέπει να γίνονται με υποδική τη ευθύνη με κάποια διάφορα διαδικασία που ε, παρέχει εγγύηση ανέξαρτησία. Νομίζω ότι αυτή τη γρεμπλέψη θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Ότι δηλαδή η Κομισιόν ήδη θα πρέπει να υποπτεύσει τι ε, διαδικασίε που εφαρμόζονται στην ιστορική τη λειτουργία. Διαβάζω τι λέει ο κ. Κάλανο όσον αφορά την προσέγγιση ΙΜΚΟ και η ΙΜΚΟ συζητά, εξετάζει τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και αποφασίζει. Οπότε, αφού εμείς έχουμε κάνει την εκτίμηση επιπτώσεων, εμείς συζητούμε μαζί σας ε, κατά αυτόν τον τρόπο την εκτίμηση επιπτώσεων. Οι εμπλεκόμενοι με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή θεώρησαν ότι αδύνατο σημείο στο σύστημα είναι ότι έχουμε τις δικές μας ε, εκτιμήσεις ε, και το θέμα είναι ποιος θα καταλάβει, ποιος μπορεί μετά να τις χτινήσει, να τις εξετάσει. Ε, όσον αφορά τώρα τι εξωτερικέ υπηρεσίε, είναι καλό παράδειγμα η υπηρεσία για το περιβάλλον, είναι εξωτερική, είναι εξάρτητη και συμμετέχει στις εκτιμήσεις επιπτώσεων και κατά ε, τον τρόπο συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Όμως δεν πρόκειται περί ενός φορέως που μπορεί να κάνει ποιοτικό έλεγχο των εσωτερικών μας εκτιμήσεων επιπτώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ja, äh, Linda, Nachfrage. Mhm. stellen, Linda. Um, Δεν ξέρω τι κάνει η ΙΜΚΟ, αλλά θέλει η Επιτροπή να μας πει πώς βλέπει την υποβολή σε εμά των εκτιμήσεων επιπτώσεων. Γιατί συνήθως γίνεται αυτή η δουλειά όσον αφορά τα δικά μας κείμενα και τις τροπολογίες. Δεν θα έπρεπε η Κομισιόν να έρχεται να μας προσθέσει ένα σημαντικό νομοθέτημα. Γιατί απορρίπτεται κάποιους τρόπους, κάποιες λύσεις και ακολουθείτε κάποιες άλλες. Ε, αυτό που μας λέτε το κάνετε και σε άλλες επιτροπές. Ε, ε, Ευχαριστώ. σχέση με αυτά που μας είπε η Κομισιόν. Η Κομισιόν έχει δική της υποδομή και φυσικά είναι σκόπιμο να τη χρησιμοποιεί για αυτές τις ε, αξιολογήσεις. Πιθανότατα οι υπηρεσίες, οργανισμοί, μπορεί αυτές να είναι αυτός ο ανεξάρτητος οργανισμός αν τους το επιτρέψουμε. Γιατί καλύτερες αρμοδιότητες από την υπηρεσία της Κοπενχάγης δεν γίνεται. Έχει μεγάλη επαγγελματικότητα και μελετάει σε πολύ ψηλό επίπεδο όλα τα προβλήματα του περιβάλλοντος σε βάθος. Και μπορούμε να την ενθαρρύνουμε να συνεργαστεί με άλλες υπηρεσίες, Φερρυπίν του Ελσίνκη για τα χημικά προϊόντα, χημικές ουσίες και με άλλες υπηρεσίες οργανισμούς για να ανταποκριθεί στην ανάγκη αξιολόγησης επιπτώσεων ανεξάρτητα και υψηλού επαγγελματικού επίπεδου. και με προαιρετική δράση εκ μέρους του Κοινοβουλίου αν αισθανθεί ότι υπάρχει ειδική ανάγκη για ορισμένα λεπτά θέματα να πάμε ακόμα ακόμα περισσότερο σε βάθος, χρησιμοποιώντας και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Αλλά επαναλαμβάνω η υπηρεσία για το περιβάλλον της Κοπεχάγης είναι άκρος επαγγελματική. Θα μπορούσαν οι υπηρεσίες οργανισμοί να πάρουν ένα ακόμα πιο ανεξάρτητο χαρακτήρα με προσθήκη κατεξαίρεση σε συγκεκριμένε περιπτώσει εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, αν υπάρξει ανάγκη. Πρόεδρο, ο κύριο Ράιτ της Κομισιόν. Θα απαντήσει. Ευχαριστώ για την πρώτη ερώτηση που θα παρουσιάσουμε και αν θα, το, παρουσιάσουμε την αξιολόγηση. Φυσικά, αν μας το ζητήσει θα το κάνουμε. Θα σας εξηγήσουμε λεπτομέρειε. για τις υπηρεσίες οργανισμού. Ναι, η υπηρεσία περιβάλλοντος είναι ανεξάρτητη, άκρος επαγγελματική. Θέτουμε ερωτήματα και ζητάμε τη γνώμη τους για την επίσης για την υπηρεσία χημικών ουσιών. Και αυτές δίνουν στοιχεία λοιπόν που περνάνε μέσα στην αξιολόγηση. Αυτό που διστάζουμε είναι η ποιότητα ελέγχου της αξιολόγησης της Κομισιόν Έχουμε δισταγμού πρώτον διότι είναι εξωτερικοί παράγοντε και δεύτερον δεν είναι ουδέτερο. Θέλουμε μια ουδέτερη αξιολόγηση. Υπάρχουν μερικέ οργανώσει επιχειρήσεων που θεωρούν ότι θα ζητηθεί και αυτόν η γνώμη. πιο καλό τρόπο να έχουμε την ουδετερότητα είναι να έχουμε όλε τι γενικέ διευθύνσει και όλου του πόλου τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Κομισιό να μελετήσουν τη μελέτη αξιολόγηση για να γίνει επαγγελματικότητα. Για να κλείσουμε ο συγγητή μα. Ευχαριστώ. Δύο σχόλια. Η διαφορά με την Κομισιόν είναι απλή. Όπως είπε και ο κύριος Ράιτ, υπάρχει ένα όργανο αξιολόγησης, ένα συμβούλιο στην Κομισιόν, απαρτίζεται από μέλη από διάφορες γενικές διαθέσεις στην Κομισιόν. Εγώ είπα αυτό το συμβούλιο να έχει και μερικά ανεξάρτητα μέλη εκτός Κομισιόν. Δέχομαι αυτά που είπε ο κύριο Ράιτ. Ε, που έχουν διαφορετικέ γενικέ διευθύνσει με διαφορετικέ προοπτικέ. Υποτίθεται να εξάρτηται. Αλλά είναι ένα μάτι από απ' έξω. Μάλλον τα δει κανεί απ' έξω. Υπάρχει υποψία η Κομισιόν να μιλάει στην Κομισιόν. Και βρίσκω ότι είναι λογικό και θα κερδίσουμε αν έχουμε και μερικού ανεξάρτητου φορεί εκτό τη Κομισιόν στο Συμβούλιο. Όχι να είναι ευρωβουλευτέ, είναι ανεξάρτητο προ τα δύο όργανα Κομισιόν και Κοινοβούλιο. Και δεύτερον, αυτά που είπε η κυρία Χάστη και άλλοι, εγώ δεν λέω να περιοριστεί η δυνατότητα των συναδέλφων να τροπολογήσουν την νομοθεσία. Και ουσιαστικά μάλιστα αυτό που λέω είναι δεν μπορούμε να επιμένουμε η Κομισιόν να μας δίνει αναλύσει, αναλύσεις κόστου-οφέλου ωφέλους και επιπτώσεων και εμείς να μην υποκείμεθα στην ίδια διαδικασία. Όχι για όλες τις τροπολογίε, αλλά για σημαντικέ τροπολογίες να είμαστε διαφανείς και ανοιχτοί όσον αφορά το κόστος μιας τέτοιας ρύθμισης. Μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να, κάνουμε πολιτική, να πάρουμε πολιτική θέση, να ξέρουμε τι κόστος έχει η κάθε πρόταση. Μπορεί να υπάρχουν και ωφέλη τη υγεία του περιβάλλοντος, κοινωνικά που είναι δύσκολο να τα εκφράσουμε με νούμερα, αλλά μπορούμε κάτι να γράψουμε δίπλα στην τροπολογία, δίπλα στην οδηγία και να κρίνουμε πολιτικά κατά πόσον αξίζει να την προωθήσουμε ή όχι. Αυτό λέω, δεν λέω να περιοριστούμε στις, στο έργο μας, να έχουμε τα στοιχεία, τα γεγονότα, τα νούμερα. Και θα περιμένω να δω τι τροπολογίες θα υποβάλουν οι συνάδελφοι στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. 15 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι στις 12 είναι προθεσμένα για την κατάθεση των Σας 13. Στις 13. Ελθόνα Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Να έρθει το απόγευμα βέβαια. Γιατί έχουμε και ενδιαφέροντα θέματα και την Προεδρία, έχουμε και την ιδέα για ένα διεθνές ε, περιβαλλοντικό ποινικό δικαστήριο, διεθνές ή ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό ποινικό δικαστήριο και για τους Γάλλους συναδέλφους Μπορείτε να κάνουμε παρέλαση στο Σαν αλλά έχουμε σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες που θα παρελάσουν μπροστά μας.